γράψω πέντε νομοθετήματα βάσει της κανονική διαδικασία του κανονισμού έχουν γίνει δεκτά αυτά τα νομοθετήματα και θα δημοσιοποιηθούν στα πρακτικά της ε, συνεδρίασης.